και ποιε δράσεις θέλει να δρομολογήσει. καλώ ήρθατε για μια ακόμη φορά και ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Okay. Excuse me. Honorable Chair. Άξια τιμή, Πρόεδρε, του μέλη της Επιτροπής. Στη ζωή είναι σημαντικό να λέμε τα πράγματα όπως έχουν, χωρίς ε, επιφυγές. Σήμερα, 26 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι χωρίς θέση εργασία. Είναι κάτι που δεν μπορούμε να το αποδεχτούμε αυτό. 7,5 εκατομμύρια νέοι Ευρωπαίοι μεταξύ 15 και 24 δεν είναι ούτε σε κάποια θέση απασχόληση ούτε σε κάποια θέση εκπαίδευση ή κατάρτιση. Αυτό δεν μπορούμε να το αποδεχτούμε και πάνω από 124 εκατομμύρια άνθρωποι είναι αντιμέτωποι με την φτώχεια ή με την κοινωνικό αποκλεισμό. Ούτε αυτό μπορούμε να το αποδεχτούμε. Γι' αυτό λοιπόν η στόχη μου για τα επόμενα πέντε χρόνια είναι απόλυτα ξεκάθαρη. Να αγωνιστούμε για πιο πολλές θέσεις εργασίας, για καλύτερη κοινωνική προστασία, και να καταπολεμήσουμε την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Αυτές είναι οι προτεραιότητες πολλών Ευρωπαίων και είμαι απόλυτα πεπισμένη ότι αυτές είναι και οι δικές σας προτεραιότητες. Αγαπητοί συνάδελφοι, ως μέλος του Κοινοβουλίου αυτού για 23 περίπου χρόνια, ο σεβασμός μου για το θεσμικό αυτό όργανο έχει αυξηθεί διαρκώς. Και δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανεί την δέσμευσή μου για μια καλύτερη Ευρώπη. Εδώ, στο Κοινοβούλιο, με λόγια αλλά και πράξει, πάντα ήθελα να υποστηρίξω την προόδο τη Ευρώπη με συγκεκριμένα αποτελέσματα όμω για τον άνθρωπο. Και αυτό πάντα το έκανα βάσει ε, πλειοψηφιών, με ευρεία υποστήριξη. Και θα ήθελα να υποδείξω ότι οι δύο τελευταίες μου εκθέσεις σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Εποπτεία και την μεταρρύθμιση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης αλλά και η δεσμευσή μου την εποχή εκείνη για να βρω μια πλειοψηφία για αυτή την οδηγία αλλά και για να υπάρξει κοινωνικός προσανατολισμός. Πάντα λοιπόν ε, λειτουργούσα πέρα από τα όρια των συνόρων, των εθνικών συνόρων, των ομάδων και πάντα σε πίστη συνεργασία με τα άλλα θεσμικά όργανα. Και αν με τη δική σας έγκριση διοριστώ ως Επίτροπος για τις απασχόλησης και κοινωνικές υποθέσεις ε, και κινητικότητα, σίγουρα θα συνεχίσω να απευθύνομαι σε αυτές τις ε, προκλήσεις. Η χρηματοπιστωτική κρίση είχε σκληρό τίμημα και τα έκτακτα μέτρα τα οποία αναγκάστηκε να πάρει η Ένωση για να καταπολεμήσει την κρίση ήταν απαραίτητα. Τώρα διαφέρονται σιγά σιγά οι θετικέ επιδράσεις ε, της πολιτικής αυτής, σιγά σιγά και αντιστακτικά. Αλλά την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων. Είναι, αυτό είναι κάτι που δεν έχουμε μπορέσει ακόμα να το πετύχουμε. Γι' αυτό λοιπόν η επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να πετύχει συγκεκριμένα αποτελέσματα τα οποία θα έχουν απτές συνέπειες για όλους τους πολίτες. Ο πρόεδρος Σαν Γιούγκερ μου ζήτησε να φροντίσω προκειμένου η λέξη κοινωνικός να ξαναποκτήσει την πλήρη σημασία της και να α, ολοκληρωθεί η οικονομία της αγοράς πλήρως. Α, αυτή την πρόκληση την αποδέχομαι γιατί είμαι πεπισμένη υποστηρίκτρια της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς όπου η ελευθερία, η υπευθυνότητα και η αλληλεγγύη συνυπάρχουν. Είναι λοιπόν σαφές ότι θα πρέπει να είναι ο στόχος μας η επόμενη επιτροπή θα πρέπει και σε κοινωνικό επίπεδο να έχει απτά αποτελέσματα από το χαρτοφυλάκιο κοινωνική, απασχόληση, κοινωνικών υποθέσεων, ικανοτήτων και εργασιακής κινητικότητας. Θέλω λοιπόν να φροντίσω να το πετύχουμε αυτό μαζί με τους ε, υποψήφιους ε, αντιπροέδρους και επιτρόπους, ιδιαίτερα με τους συναδέλφους ο Νομπροβόσκη και Μοσκοβίτση, θα δουλέψουμε ως μία ομάδα και θεωρώ ότι θα είναι δική μου, δικό μου καθήκον προκειμένου να φροντίσουμε τα επόμενα πέντε χρόνια η πολιτική σε όλους τους τομείς να λάβει υπόψη όλες τις κοινωνικές επιπτώσεις των μέτρων. Όπως είπε ήδη ο Jean-Claude Juncker, δεν θα έχουμε εξέλθει από την κρίση όσο 26 εκατομμύρια συμπολιτών μας εξακολουθούν να παραμένουν άνεργοι. Κατά τη γνώμη μου δεν θα πρέπει να κάνουμε μια επιλογή μεταξύ ανταγωνιστικότητας και κοινωνικής ισότητας. Πρόκειται για τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος που από κοινού αποτελούν το βάθρο της ε, κοινωνικής οικονομίας της αγοράς που είναι ανταγωνιστική και αλληλέγγυα. Ο ρόλος μου θα είναι να συμβάλλω στη διαμόρφωση των καλύτερων προϋποθέσεων για να επιστρέψουν οι άνεργοι στην αγορά εργασίας και να καταπολεμήσουμε τον κοινωνικό αποκλεισμό και τη φτώχεια. Αυτό προϋποθέτει την ανάπτυξη μιας αγοράς εργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μιας αγοράς εργασίας που θα είναι δυναμική και ολοκληρωμένη. Εκεί που οι ετούντες θέσεις απασχόλησης θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες και προσόντα για να ανταποκριθούν στις ανάγκες των επιχειρήσεων όπου και αν βρίσκονται αυτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση μία κατάρτιση που θα πρέπει να είναι προσιτή σε όλους, να είναι προσαρμοσμένη σε ανάγκες, να επικεντρώνεται ιδιαίτερα στους μακροχρόνια άνεργους και στην κινητικότητα των εργαζομένων. Όλα αυτά είναι απαραίτητα μέτρα σήμερα για την Ευρώπη για να ξαναβρούμε το δρόμο της οικονομικής ανάπτυξης και να μειώσουμε τη φτώχεια. Όσες και όσοι με γνωρίζουν, γνωρίζουν κάλλιστα ότι δεν ψάχνω ποτέ απλοϊκές λύσεις για περίπλοκα προβλήματα. Κάτι τέτοιο δεν είναι ούτε αξιόπιστο, ούτε έντιμο, αλλά ούτε και αποτελεσματικό. Θέλω απτά αποτελέσματα. Θέλω οι επιχειρήσεις να αναπτύσσονται και να προσαρμόζονται στις ραγδαίες εξελίξεις της παγκοσμιοποίησης, στην οποία συμμετέχουμε ενεργά. Θέλω ταυτόχρονα εργαζόμενοι και εργοδότες να συμβάλλουν με την εργασία τους στην δημιουργία πλούτου με προϋποθέσεις όμως που θα εξασφαλίζουν την αξιοπρέπειά τους, τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους και την ισότητα των ευκαιριών. Άνδρες και γυναίκες, υπήκοοι της χώρας στην οποία απασχολούνται ή άλλης χώρας, ανάπηροι, όλοι πρέπει να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας και όλοι έχουν δικαίωμα και αξίζουν ίση αμοιβή για ίσες υπηρεσίες, για ίση εργασία. Εξάλλου, η διαφύλαξη της ανταγωνιστικότητάς μας και η διαχρονικότητα των κοινωνικών συστημάτων προστασίας μας απαιτούν την, τον εντοπισμό των καταχρήσεων και την ε, τιμωρία τους. Γι' αυτό θα ε, δώσω έμφαση σε τέσσερις προτεραιότητες που έχουν ίση σημασία και αυτές θα προσπίσω. Καταρχήν, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Πολλές θέσεις εργασίας ε, έχουν καταστραφεί, καταρακωθεί από την κρίση. Εκατομμύρια. Για να δώσουμε λοιπόν νέες προοπτικές στους ανέργους, θα πρέπει να δημιουργήσουμε νέες θέσεις απασχόλησης. Οι επιχειρήσεις και κυρίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρειάζονται ευνοϊκές ε, συνθήκες για να ξεκινήσουν και να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους, είτε παραδοσιακές είτε καινοτόμες, και να κατακτήσουν νέες αγορές. Δεύτερον, πρόσβαση στην απασχόληση. Μία μαζική απασχόληση συνυπάρχει με ένα γεράσκον εργατικό δυναμικό και, και με ανέργους, κυρίως νέους, που συχνά είναι ανειδίκευτοι, δεν έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες και δεν έχουν πια πρόσβαση σε σταθερές ε, θέσεις εργασίας. Χρειαζόμαστε λοιπόν περαιτέρω προσπάθειες για να καθοδηγήσουμε και να προσανατολίσουμε τους νέους και να επιτρέψουμε στις γυναίκες και στους αναπήρους πλήρη πρόσβαση στην αγορά εργασίας και επίσης να επανενεργοποιήσουμε τους μακροχρόνια άνεργους. Μεταξύ των λύσεων που προτείνω είναι μια καλύτερη κινητικότητα των εργαζομένων. Θα πρέπει λοιπόν αυτή την κινητικότητα να την προωθήσουμε. Τρίτον, δεξιότητες, προσόντα. Η ανταγωνιστικότητά μας εξαρτάται πρώτα απ' όλα από τις δεξιότητές μας. Οι εργαζόμενοι σήμερα στη διάρκεια του ενεργού τους βίου έχουν πολλές επαγγελματικές σταδιοδρομίες. Θέλουμε λοιπόν να καλύψουμε τις καθυστερείς τους και τα κενά τους στην ε, απόκτηση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων και προσόντων ε, για τους εργοδότες και τους εργαζόμενους ασχέτως της ηλικία τους. Τέταρτον, η κοινωνική προστασία. Η κοινωνική προστασία είναι θεμελιώδης επένδυση και βάση της ε, ευημερία μας. Το 2010 διατυπώσαμε ένα ξεκάθαρο στόχο, ότι μέχρι το 2020 θέλουμε να μειώσουμε κατά 20 εκατομμύρια τον αριθμό των ανθρώπων που είναι θύματα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Δυστυχώς το αντίθετο συνέβη. Η κρίση οδήγησε σε μια απότομη αύξηση της φτώχειας και του αποκλεισμού. Τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας που έχουμε θα πρέπει να είναι πιο αποτελεσματικά και καλύτερα προσανατολισμένα στα αποτελέσματα, διασφαλίζοντας μια ειφορία μακροπρόθεσμα. Αγαπητοί συνάδελφοι, για να υλοποιήσουμε τις προτεραιότητες αυτές θα χρησιμοποιήσω όλα τα μέτρα και τους μηχανισμούς που έχω στη διάθεσή μου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα επικεντρωθώ κυρίως σε τέσσερις άξονες. Πρώτον, κινητοποίηση των απαραίτητων επενδύσεων. Στόχος μου είναι να προωθήσω τις επενδύσεις για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και να βοηθήσω στην επαναφορά των ανέργων στην αγορά εργασία. Γι' αυτό και θα συνεργαστώ με τον Αντιπρόεδρο Γύρ Κατάινεν για να ετοιμάσουμε την κινητοποίηση 300 δισεκατομμυρίων ευρώ επενδύσεων που έχει αναγγείλει ο Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ. Σα διαβεβαιώ ότι θα κινητοποιήσω όλα τα διαθέσιμα χρηματοπιστωτικά εργαλεία και μηχανισμούς για να επενδύσω στους ανθρώπους, ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Ευρωπαϊκής Ενίσχυσης στους Απόρους και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Όλα αυτά τα ταμεία και τα κονδύλια τους θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία θέσεων απασχόληση, δημιουργία δεξιοτήτων και καταπολέμηση της φτώχειας. Επίσης, θα επιταχύνω την εφαρμογή της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων στα κράτη-μέλη. Και γι' αυτό θα πρέπει να δώσουμε σάρκα και οστά στο, στα προγράμματα για την εγγύηση για την νεολαία. Δεύτερον, η οικονομική διακυβέρνηση θα πρέπει να αλλάξει ταχύτητα. Η απασχόληση και οι κοινωνικέ πολιτικέ θα πρέπει να είναι πιο παρούσε στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Θα συνεργαστώ λοιπόν στενά με τον Αντιπρόεδρο Βάλτη Ντομπρόφσκη και τον συνάδελφο Μοσκοβισή, ώστε οι αποφάσεις που λαμβάνουμε να λαμβάνουν καλύτερα υπόψη τις κοινωνικές επιπτώσεις των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Η ευάθυνση των μεταρρυθμίσεων στα κράτη-μέλη είναι απαραίτητη, αλλά κάτι τέτοιο προϋποθέτει μεγαλύτερη δικαιοσύνη και βιωσιμότητα των μεταρρυθμίσεων. Ο κοινωνικός αντίκτυπος ε, των ε, προγραμμάτων διάσωσης για έφευσες χώρες θα πρέπει να συμβάλλουν σε αυτό το στόχο. Επίσης θα πρέπει να επενεκκινήσουμε τον κοινωνικό διάλογο. Θα συνεργαστώ με τον Αντιπρόεδρο τον ώστε οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο να γίνουν πραγματικοί εταίροι μας στο ευρωπαϊκό εξάμεινο. Οι σημαντικές και δύσκολες κοινωνικές μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να συζητηθούν πλήρως με τους κοινωνικούς εταίρους και να εμπλέκουν όλους τους βασικούς φορείς ε, και να καλύπτουν όλο το οικονομικό και κοινωνικό φάσμα συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενων που αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των θέσεων απασχόλησης στην Ευρώπη σήμερα. Τρίτον, αναλογικότητα στους κοινούς κανόνες. Έτσι θα δημιουργήσουμε συνθήκες ίσου ανταγωνισμού και θα προασπίσουμε την ενιαία αγορά χωρίς να δημιουργούμε υπερβολικό άχθος για τους διάφορους φορείς. Θα συνεργαστώ στενά με τα κράτη-μέλη για να εξασφαλίσω μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Αυτό το σημείο θα πρέπει να ενισχυθεί. Και σύμφωνα με, την, με το πρόγραμμα για την έξυπνη νομοθεσία, θα αξιολογήσω την υφιστάμενη νομοθεσία προκειμένου να είναι αποτελεσματική, αναλογική και εύχρηστη, εύκολης εφαρμογής. Θα πρέπει επίσης να προστατεύσουμε τους εργαζόμενους από νέους κινδύνους και γι' αυτό θα προτείνω τον εξυγχρονισμό και όπου δει και την απλούστευση του νομοθετικού μας κεκτημένου ενώ ταυτόχρονα θα διασφαλίσω ένα υψηλό επίπεδο προστασίας. Θα εξετάσω και θα υποβάλω και νέες πρωτοβουλίες όπου χρειάζεται, για παράδειγμα στο θέμα της κινητικότητας των εργαζομένων. Τέλος, καθήκον μου είναι να αξιοποιήσω στο έπακρο τους μηχανισμούς και τις εταιρικέ σχέσεις που έχουμε και τα επόμενα χρόνια από κοινού και σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη, με τους κοινωνικούς εταίρους και τους συναδέλφους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να δημιουργήσουμε μια Ευρώπη πιο δίκαιη και πιο βιώσιμη. Την επόμενη πενταετία θα έχω στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα είμαι στη διάθεσή σας για να συζητούμε τακτικά την πορεία των εργασιών μας. Έχουμε ένα κοινό στόχο. Τους ανθρώπους, την υγεία τους, την δουλειά τους, την ευμάρειά τους. Η Ευρώπη είναι για τους ανθρώπους και μπορείτε να υπολογίζετε σε μένα. Θα είμαι ο σύμμαχός σας για να πραγματώσουμε αυτό το στόχο. Ευχαριστώ.